Euh, Αγαπητοί συνάδελφοι, αν συμφωνείτε να αρχίσουμε τη συνεδρία της Επιτροπής μας. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε σήμερα το απόγευμα τη συνέχεια της εργασίας της ε, Επιτροπής ε, Ανάπτυξης μετά την συζήτηση που είχαμε για τα θέματα φίλου με την Επιτροπή ε, Δικαιωμάτων των Γυναικών. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι εγκρίνεται η μέρη στη διάταξη που έχετε στο φάκελό σα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στο σημείο 3. Να υπενθυμίσω ότι την προσεχή Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου, στο Στρασβούργο, στις 7.30 το απόγευμα, θα έχουμε κοινή συνεδρίαση AFEDE όπου θα παρουσιάσουμε τις έξι προτάσεις για την απονομή του βραβείου Ζαχάροφ 2017. Το επενθυμίζω γιατί άλλαξε η ημερομηνία και ο χώρος της συνεδρίασης. Η συνεδρίαση θα γίνει και η ώρα άλλαξε. Στην αίθουσα λοιπόν θα γίνει συνεδρίαση low N14 στο Στρασβούργο. 4. Έγκριση των αποφάσεων και συστάσεων των συντονιστών που ελήφθησαν στις 6 Σεπτεμβρίου και υπάρχουν στο φάκελό σας. Αν έχετε παρατηρήσεις, παρακαλώ να ενημερώσετε τη γραμματεία πριν το τέλος της συνεδρίασής μας. Εάν δεν υπάρξουν παρατηρήσεις, θα θεωρηθεί ότι οι αποφάσεις των συντονιστών της 6 Σεπτεμβρίου ενεκρίθησαν. Σημείο 5. Ανακοινώσει Επιτροπής. Θα ήθελε να μας ενημερώσει η Επιτροπή για κάποια θέματα. Ωραία. Α, όχι. Καλώς. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα περνάμε στο σημείο 6 της ημερήσιας διάταξής μας. Νέα όργανα και βέλτιστες πρακτικές για την ανθρωπιστική βοήθεια, ιδιαίτερα στα πλαίσια των ε, μετατοπισμένων ε, μακροχρόνιας διάρκειας. Το σημείο αυτό είναι μια ανταλλαγή απόψεων για τις βέλτιστες πρακτικές και τα νέα εργαλεία, ιδιαίτερα στα πλαίσια μακροχρόνιας μετατόπισης. Ξέρουμε όλοι ότι η ανθρωπιστική βοήθεια αντιμετωπίζει όλο και περισσότερες κρίσεις ε, που διαρκούν όλο και περισσότερο λόγω θεομηνιών ή ε, προβλημάτων από τη δράση των ανθρώπων. Γι' αυτό είναι όλο και πιο πιεστικές οι ανάγκες και πρέπει με περιορισμένους πόρους να αντιμετωπίσουμε όλο και περισσότερες καταστάσεις τα τελευταία χρόνια. Έχουμε συζητήσει για τους τρόπους μεταρρύθμισης του συστήματος ανθρωπιστικής βοήθειας για να γίνει πιο αποτελεσματικό. Η οργάνωση της ε, πρώτης συνάντησης κορυφής για ανθρωπιστικά θέματα στην Κωνσταντινούπολη τον Μάιο, Μάιο του 2016 και η ολοκλήρωση της ε, διαπραγμάτευσης μεταξύ των ε, κυριωτέρων δωρητών και τους κυριότερους οργανισμούς παροχής της βοήθειας είναι συγκεκριμένα παραδείγματα αυτών των συζητήσεων. Μία από τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στα πλαίσια αυτής της ε, μεγάλης διαπραγμάτευσης είναι να βασιστούμε στην ε, παροχή ε, χρηματικής βοήθειας στα πλαίσια της ανθρωπιστικής βοήθειας. Η παροχή χρηματικής βοήθειας, δηλαδή σε μετρητά, βοηθάει να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά οι ανάγκες και να γίνουν ευκολότερα και οι εμπορικές συναλλαγές. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό στα πλαίσια των μακροχρονίων κρίσεων που σχετίζονται με την μετατόπιση πληθυσμών. Μέχρι πρόσφατα οι παροχές ε, βοήθειας μετρητών ήταν περιορισμένες. Αλλά σε κάθε πλαίσιο κρίσης η κατάσταση είναι διαφορετική και αξιοποιώντας τις διάφορες καταστάσεις μπορέσαμε να επεκτείνουμε την ε, παροχή μετρητών τα τελευταία χρόνια. Για να συζητήσουμε την παροχή βοήθειας μετρητά, σε μετρητά έχουμε δύο διακεκριμένους εμπειρογνώμενες, την κυρία Χενρίκε Τραουτμάν που είναι τμήματάρχης για την ε, πολιτική για την ανάπτυξη και την περιφερειακή στρατηγική στην Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ και την κυρία Δάφνη Γιαγιασίνκε που είναι κύριος σύμβουλος για τα θέματα οικονομικών προγραμμάτων στα πλαίσια της Διεθνούς Οργάνωσης ε, Παροχής Βοήθειας και Διάσωσης. Η κυρία Τράτμαν θα μας ενημερώσει για τις συζητήσεις που γίνονται στους διεθνείς οργανισμούς στα πλαίσια της εφαρμογής αυτής της μεγάλης διαπραγμάτευσης. Και η κυρία Γιασιγκέ θα συμπληρώσει αυτή την παρουσίαση με μια αναλυτική παρουσίαση των ε, λεπτομεριών οργάνωσης της παροχής αυτών των ε, βοηθειών σε μετρητά στα πλαίσια των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων διάσωση. Να δώσω λοιπόν το λόγο στις εμπειρογνώμονές μας, όταν πόνε η κυρία Τροτμάν. 10 έως 15 λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, κύριε και κύριοι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας για να σας κάνουμε μια επισκόπηση τι γίνεται για την παροχή βοήθειας σε μετρητά και τις γενικότερες εξελίξεις ε, στην αντιμετώπιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα σας δείξω καταρχάς ένα σύντομο βίντεο για να καταλάβετε τι γίνεται και μετά θα επανέλθω. Humanitarian crises, be they due to conflict or natural disasters, are affecting increasing numbers of people. In order to meet the needs of those affected by crisis,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 Νομίζω ότι καταλάβατε πολύ καλύτερα από ό,τι θα μπορούσα να σα εξηγήσω, αλλά να περάσω μερικά βασικά θέματα. Η χορήγηση μετρητών είναι αποτελεσματικό τρόπο για τη χορήγηση ανθρωπιστική βοήθεια σε πολλά πλαίσια, όχι σε όλα, αλλά σε πολλά. Μα δίνει περισσότερη αξιοπρέπεια, επιλογή και ευελιξία. Και είναι η καλύτερη χρήση των χρημάτων και για του δωρητέ και για του ε, φορολογούμενου. Επίση υποχρεώνει τις ε, ανθρωπιστικές οργανώσεις επιτόπου να συνεργαστούν περισσότερο. Και πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένη η παροχή βοήθεια σε χρήματα. Δεν μπορεί να γίνεται με τον ίδιο τρόπο στο Λίβανο όπω στη Σομαλία, αλλά μπορεί να γίνει σχεδόν παντού, κατά τη γνώμη μα. Επίση, έτσι τίθεται ένα αμφιβόλο η παραδοσιακή ανθρωπιστική βοήθεια που γίνεται κατά τομέα, για παράδειγμα τρόφιμα, φάρμακα κτλ μας ε, υποχρεώνει να αντιμετωπίσουμε σφαιρικά το θέμα. Γι' αυτό θεωρούμε ότι θα πρέπει να αυξηθούν οι προσπάθειες παροχής βοήθειας σε μετρητά που είναι κάτω από 10%. Η γενική μου διεύθυνση το 2016 ήδη έχει χορηγήσει το 33% της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης σε όλους τους τομείς σε μετρητά. Κυρίως ε, χορηγείται για την ε, αγορά βοήθειας, ε, ενώ η στέγαση και άλλες υπηρεσίες που ονομάζονται WASH ε, εξακολουθούν να είναι σε μικρότερο βαθμό. Ιδιαίτερα όταν υπάρξει ανάγκη άμεσης αντίδρασης. Δεν χρειάζεται λοιπόν να χορηγηθούν μέσω αεροπορικής μεταφοράς κάποια βοήθεια. Και είναι λοιπόν πάνω από 54% 16%. Η μεγάλη διαπραγμάτευση που ήδη αναφέρθηκε, τι λέει για την χορήγηση μετρητών. Όσοι έχουν παρακολουθήσει τη συζήτηση γνωρίζουν ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία για τη χορήγηση βοήθεια σε χρήματα για να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο τα προγράμματα αυτά αλλά δεν συμφωνήθηκε ο στόχος και ορισμένοι δωρητές έχουν καθορίσει συγκεκριμένους στόχους μόνοι τους, μονομερός. Η γενική μας διεύθυνση θέλει μέχρι το τέλος του 17-35% της βοήθειας να δίδεται σε μετρητά και με τάση αυξητική περαιτέρω. Επίσης θέλουμε να παρακολουθούμε και να αξιολογούμε την ε, χορήγηση βοήθειας σε μετρητά. Γιατί έτσι μας επιτρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια να αξιολογήσουμε αν είναι καλύτερο αυτό το σύστημα. Και πρέπει να συλλέξουμε στοιχεία Έχουμε πολλά στοιχεία, αλλά πάντα μπορούμε να συλλέξουμε και να τα αξιοποιήσουμε καλύτερα και αυτό προσπαθούμε τώρα. Και τι στοιχεία έχουμε μέχρι στιγμής. Θα υπάρξει μια έκθεση από το 2015 μια ομάδα εργασία υψηλού επίπεδου που κοίταξε όλα τα αποτελέσματα τη έρευνα και τις λεπτομέρειες, αλλά θα συνοψίσω. Η χορήγηση μετρητών είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική σε μεγάλη κλίμακα, δηλαδή όταν υπάρχει μια κρίσιμη μάζα γι' αυτό αν έχετε 22 διαφορετικούς οργανισμούς που παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια και όλοι δίνουν ε, ένα μικρό ποσοστό της βοήθειάς τους σε χρήματα, δεν καταλήγει σε αυτή την κρίσιμη μάζα. Πρέπει να γίνεται μέσω μιας συγκεντρωτικής μεγάλης προσπάθειας. Όπως κάνουμε τώρα στη Μέση Ανατολή, στο Λίβανο. Και επίσης ε, τα μετρητά ε, τονώνουν τη λειτουργία των αγορών. Το λέει και το βίντεο, αλλά υπάρχει σαφής ε, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι γίνεται αυτό. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Οι κίνδυνοι που φοβόμασταν δεν προέκυψαν. Πολλοί ανησυχούσαν ότι όλα αυτά θα δαπανώνται σε τσιγάρα, ναρκωτικά, ενόπνευμα. Και ξέρουμε ότι αυτό προέκυψε πριν από δύο χρόνια κατά την κρίση. Ε, προέκυψε δηλαδή ε, να, ο φόβος ότι θα μπορούσαν να πληρώνονται μέσω αυτής της βοήθειας και οι διακινητές, αλλά δεν προέκυψε. Ιδιαίτερα αν παρακολουθείτε σωστά η χρήση της βοήθειας σε μετρητά. Και η χορήγηση μετρητών αποδεικνύει ότι περισσότερη βοήθεια φτάνει στους δικαιούχους και μειώνει και τις απώλειες λόγω της περαιτέρω πώληση, της μεταπώλησης της παραδοσιακής ανθρωπιστικής βοήθειας. Υπάρχει μια συγκεκριμένη έκθεση που δείχνει ότι το σόργο και η ζάχαρη και το ρύζι ε, μεταπολούνται μετά σε κάποιους που ήδη περιμένουν. Γιατί χορηγείται βοήθεια που, που ενδεχομένως δεν τη χρειάζονται οι δικαιούχοι. Αυτό σταματάει έτσι. Δεν χάνεται ένα τμήμα της αξίας της βοήθειάς μας μέσω μεταπόληση. Και πολύ συχνά είναι ένα πρώτο βήμα για να αρθεί ο οικονομικός αποκλεισμός ε, των ατόμων που δικαιούνται, που επωφελούνται. Αποφασίζουν πώς θα αξιοποιήσουν αυτή τη χρηματική βοήθεια αλλά αναπτύχθηκε αυτός ο τρόπος βοήθειας τόσο γρήγορα αυτά τα δύο τελευταία χρόνια που εμείς ως Επιτροπή θεωρούμε ότι πρέπει να δώσουμε περισσότερη βοήθεια στους ε, δικαιούχους και στους οργανισμούς που παρέχουν τη βοήθεια. Όπως κάνουμε τώρα στο Λίβανο, στην Ιορδανία και την Τουρκία. Είναι τουλάχιστον 2 εκατομμύρια ευρώ σε καταστάσεις σταθερές και προστατευόμενες όπου είναι πάνω κάτω σταθερές οι καταστάσεις, σταθερός ο αριθμός των μετατοπισμένων. Δεν χρειάζεται κάθε δύο μήνες, αν ε, μετατοπιστούν περαιτέρω τα άτομα, όπως το Λίβανο δηλαδή, που δεν μετατοπίζονται, να ξαναδείς όλο το σύστημα. Κάποιες θα πρέπει να είναι αρχές. Πρώτα απ' όλα πρέπει να έχει αποτελεσματικότητα. Θέλουμε ένα ενιαίο σύστημα παράδοσης ε, των μετρητών και ένα σωστό ε, λόγο μεταξύ των πιστώσεων που χορηγούμε και των πιστώσεων που φτάνουν στους δικαιούχους. Ε, αν δεν ξέρουμε τι ποσοστό δίδεται από ένα δωρητή σε έναν οργανισμό του ΟΗΕ, σε μια τοπική μη κάπα όμικρον και τελικά στο δικαιούχο, αν δεν ξέρεις τι ποσοστό χάνεται στο δρόμο, γιατί έχουμε στοιχεία που λένε ότι μπορεί και 50% να χάνεται στο δρόμο. Ε, αν δεν έχει λοιπόν ένα τέτοιο ε, ποσοστό, ένα καλό ποσοστό που να φτάνει, και δεν λέω ότι όλα όσα χάνονται, χάνονται άσκοπα και τόσε φορές τίθενται θέματα ασφάλειας και άλλα έξοδα. Αλλά το βασικό είναι το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό της βοήθειας να φτάνει στους δικαιώχους. Με μετρητά θεωρούμε ότι έχουμε πολύ καλύτερο λόγο, καλύτερο ποσοστό για την Τουρκία για παράδειγμα. Δηλαδή θεωρούμε στην Τουρκία ότι το 85% των πιστώσεων φτάνει στο δικαιούχο και μόνο 15 χάνεται στο δρόμο. Και μπορούμε, πιστεύω, εάν ε, εστιάσουμε περισσότερο σε μετρητά, να αυξήσουμε αυτό το ποσοστό. Επίση, θα πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα παράδοση, όχι 22 διαφορετικέ οργανώσει με διαφορετικέ ε, τραπεζικέ κάρτε, χρεωστικέ κάρτε, ένα να ασχολείται με το WOS, άλλο με τη διατροφή, άλλοι με την προστασία κτλ. Να υπάρχει σταθερό αριθμό δικαιούχων, σταθερό πλαίσιο για να καλύπτονται όλοι με τον ίδιο τρόπο και να υπάρχει και αναγκαία κρίσιμη μάζα και οικονομίες μεγέθους. Γι' αυτό θέλουμε να υπάρχουν δύο στοιχεία. Από τη μία ανθρωπιστική επιχείρηση και από την άλλη οι μεταφορές μετρητών. Αυτό θα μας επιτρέψει να έχουμε περισσότερη διαφάνεια, ιδιαίτερα για το τι στοιχεία κόστους προκύπτουν και ε, καλύτερη λογοδοσία και στις δύο πλευρές, και τους δωρητές και τους ε, δικαιούχους ε, στο Λίβανο για παράδειγμα μπορούμε να συνδέσουμε αυτές τις ε, πληρωμές και με τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας υποδοχής δεν χρειάζεται να δημιουργήσουμε ένα παράλληλο σύστημα. Εάν το κράτος υποδοχής τους επιτρέπει να παραμείνουν μπορούμε να αξιοποιήσουμε και τα τοπικά συστήματα κοινωνικής πρόνοιας για να λάβουν την αναγκαία βοήθεια. Το θέμα δεν είναι να τους δίνεις μόνο κουβέρτες και καύσιμα, είναι να τους δίνεις δυνατότητα να δημιουργήσουν μια ζωή. Διατηρούνται οι, τα άλλα συστατικά, θα υπάρχει προστασία, θα υπάρχει στόχευση και παρακολούθηση των αδυναμιών και θα μπορούμε πάντα να επανέλθουμε σε ένα πιο παραδοσιακό σύστημα βοήθεια σε είδο, αν δεν λειτουργούν οι αγορέ, αν υπάρχει συνεχής μετατόπιση, αν υπάρξει μαζική ε, άφηξη ατόμων. Αλλά γενικά ε, η μακροπρόθεσμη προοπτική μας είναι να εδραιωθούν οι πληρωμές σε μετρητά. Νομίζω ότι υπήρξε λοιπόν βασική αλλαγή προσέγγισης. Είναι κάτι καινούριο λοιπόν αυτό το σύστημα. Δεν το έχουμε κάνει μέχρι τώρα το να έχουμε μόνο ένα σύστημα παράδοσης ε, και ε, έναν οργανισμό παράδοσης μας επιτρέπει περισσότερο συντονισμό. Για να το επιτύχουμε αυτό βέβαια πρέπει να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις, αλλά μας δίνει οικονομίες κλίμακος και έχει αποτελέσματα επιτόπου. Και θα συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε και τις άλλες πλευρές αυτοί λοιπόν οι κανόνες για την ε, χορήγηση μετρητών σε μεγάλη κλίμακα. Αλλάζει ιδιαίτερα έτσι και ο τρόπος λειτουργίας ε, των υπηρεσιών μας. Συνεχίζουμε όπως να λειτουργούμε και με τους παραδοσιακούς μας εταίρους. Θα μπορούσαμε για παράδειγμα να εντάξουμε και ιδιωτικές επιχειρήσεις που θα ασχοληθούν μόνο με την ε, τελική πράξη χορήγησης των χρημάτων μέσω μιας εταιρεία ε, πιστοτικών καρτών, για παράδειγμα, Mastercard. Κάτι που θα μας επέτρεπε να ασχοληθούμε κυρίως με τα ανθρωπιστικά μα καθήκοντα και να μην ασχολούμεθα με θέματα που είναι χρηματοοικονομικής φύσης. Δεν λέω ότι μπορεί να γίνει ήδη αυτό, αλλά πρέπει να αρχίσουμε να το εξετάζουμε και όχι απλώς να τις αναφέρουμε. Έτσι μπορούμε να ε, εμπλέξουμε περισσότερο και τους ίδιους τους δικαιούχους και τους εκπροσώπους τους. Ο συντονισμός των δωρητών είναι επίσης πολύ σημαντικότερος, γιατί ξέρετε ότι οι διάφοροι δωρητές ε, χρηματοδοτούν ε, διάφορες πλευρές της βοήθειας χωρίς να συνομιλούν μεταξύ τους, άρα το βασικό είναι να υπάρχει η καλύτερη κρίσιμη μάζα, για να έχει την καλύτερη, το καλύτερο αντίκτυπο. Αυτές οι πληρωμές μετρητά μας επιτρέπουν να βελτιώσουμε όπω το Λίβανο την κατάσταση. Είχαμε πολύ θετικέ εμπειρίες εκεί η βοήθεια που δίδει η Γερμανία, η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση συντονίζονται μεταξύ τους και βοηθούν να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Τώρα η διευκόλυνση για την Τουρκία. Νομίζω ότι εκεί έχουμε ήδη ένα ενίο σύστημα παροχής που χρηματοδοτείται μέσω του WFP δεν χωρίς συνθήκες ε, τα μετρητά, αλλά έχουμε και άλλες ε, χρηματοδοτήσεις σε είδος, όπου η χρηματοδότηση ε, στοχεύει κάποια συγκεκριμένη βοήθεια, για παράδειγμα εκπαίδευση. Λέμε ότι πρέπει να δοθούν αυτοί οι πόροι για την εκπαίδευση των παιδιών σας για να μην αποκλειθούν εντελώς από το σχολικό σύστημα. Υπάρχει συντονισμός των διαφόρων κυβερνητικών και μη κυβερνητικών εταίρων. Και εμείς που είμαστε δωρητές έχουμε και μία στρατηγική εξόδου. Γιατί το σύστημά μας η SSN σχετίζεται με το σύστημα κοινωνικής προστασίας μπορούμε να εντάξουμε τη βοήθειά μας στην αναπτυξιακή βοήθεια που ε, είναι αντικείμενο διαχείρισης από άλλη υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έτσι έχουμε περισσότερη διαφάνεια η ανταλλαγή πληροφόρησης γίνεται με πολύ πιο ρευστό τρόπο και ε, μπορούμε πολύ πιο ενεργά να εντάξουμε την προσπάθεια αυτή στην κοινωνία. Στατιστικά στοιχεία. Στην αρχή είχαμε 4.000 δικαιού, δικαιούχους, στο τέλος του 2016, μόνο δηλαδή πριν από 9 μήνες και πιστεύω ότι σε δύο εβδομάδες θα ξεπεράσουμε το εκατομμύριο και θα φτάσουμε στα 1,3 μέχρι τέλος του χρόνου. Είναι περίπου το 1 τρίτο λοιπόν των εγγεγραμμένων προσφύγων στην Τουρκία και αν συνεχιστεί αυτή η διευκόλυνση θα αυξηθεί και ο αριθμός δικαιούχων. Έχουμε ήδη ε, καταβάλει το αρχικό κόστος εγκατάστασης του συστήματος και πιστεύω ότι πάνω από 50% των περαιτέρω χρηματοδοτήσεων θα φτάνουν στους δικαιούχους. Τέλος. Ε, μετρητά και τεχνολογία. Πολύ σημαντικό. Δεν θα ήταν δυνατόν να υλοποιήσουμε αυτές τις αλλαγές χωρίς ε, την αξιοποίηση των ε, τεράστιων αλλαγών στην τεχνολογία. Για παράδειγμα, οι συνδρομές στην κινητή τηλεφωνία μεταξύ του 2000 και του 2012 έχουν αυξηθεί κατά 2.500%. Στην Κένια, για παράδειγμα, 30% του ΑΕΠ διακινείται μέσω ε, μεταφορών μέσω κινητών τηλεφώνων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για όσου μπλέκονται στην προσπάθεια ανθρωπιστική βοήθεια. Θα δείτε σε μερικέ διαφάνειε Αυτές οι μεταφορές χρημάτων δίδονται μέσω, γίνονται μέσω κινητής τηλεφωνίας, χωρίς δηλαδή χαρτονομίσματα σε φακέλους, αλλά αυτό δίνει και στις γυναίκες τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην οικονομική ζωή γιατί παίρνουν ε, τα χρήματα απευθείας στο κινητό και αποφασίζουν πώς να τα δαπανίσουν. Και μέσω των κινητών είναι και πιο ασφαλείς οι ε, δοσοληψίες η χρήση βιομετρικών στοιχείων ε, βοηθάει να καταπολεμήσουμε τις απάτες. Διασφαλίζουμε έτσι ότι τα χρήματα φτάνουν στους πιο ευάλωτους. Και οι νέες εξελίξεις, το blockchain, η κρυπτογράφηση, θα μας πάρουν κανένα δύο χρόνια ακόμη, αλλά πιστεύουμε ότι θα αξιοποιηθούν. Είναι λοιπόν πολύ πιο απλή η κατάσταση, αλλά χρειάζεται διαλειτουργικότητα των συστημάτων και τρόπους ακριβώς επικοινωνίας μεταξύ των συστημάτων, δηλαδή η ψηφιακή ταυτότητα, όλα αυτά υπερβαίνουν την ε, σημερινή μας συνάντηση, αλλά είναι πολύ σημαντικά για τον ανθρωπιστικό τομέα, δηλαδή όλοι κάποια στιγμή θα μπορούν να αναγνωρίζονται μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας ανεξάρτητα από το σε ποια χώρα μετακινούνται. Αυτό θα το παρακολουθήσουμε. Βεβαίως ε, αυτές οι δοσοληψίες σε μετρητά, διαταράσσουν την παραδοσιακή ανθρωπιστική παροχή βοήθειας. Σε ορισμένα μέρη δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει γιατί δεν υπάρχει η τεχνολογία, δεν υπάρχει η ασφάλεια, δεν υπάρχουν τα συστήματα κοινωνικής προστασίας, αλλά υπάρχουν δυνατότητε περαιτέρω διεύρυνσης αυτών των δυνατοτήτων. Πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα βγει από μια στενή αντιμετώπιση, ανθρωπιστική βοήθεια, όπου ο καθένα δουλεύει στη γωνίτσα του χωρίς να συνομιλεί με τους άλλους. Μέσω των μετρητών μπορούμε να στοχεύσουμε καλύτερα τις ανάγκες των δικαιούχων και να τις καλύψουμε μέσω πληρωμών σε μετρητά. Θεωρούμε ότι έτσι μπορούμε να βοηθήσουμε αυτούς που έχουν θυγεί από τις κρίσεις να έχουν περισσότερη επιλογή και την εμπλοκή και ιδιωτικών φορέων και επιχειρήσεων. Όπως είπα και στην αρχή, έχουμε τόσο πολλές κρίσεις στον κόσμο, όλα κοστίζουν περισσότερο, αλλά δεν αυξάνονται οι προπολογισμοί μας. Προσπαθούμε λοιπόν και με τη δική σας βοήθεια να κάνουμε ό,τι μπορούμε, δεν τα καταφέρουμε πάντα, αλλά θα πρέπει να έχουμε καλύτερη απόδοση για τις πιστώσεις μας. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπετε εδώ και κάποια link για περαιτέρω ενημέρωση και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστώ την κυρία Τρότμαν. Η κυρία Γιαγιά Σίγκε τώρα για 10 με 15 λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και την Επιτροπή Ανάπτυξης που προσκάλεσε τη Διεθνή Επιτροπή Διάσωσης. Η Διεθνή Επιτροπή Διάσωσης ε, έρχεται να δώσει απαντήσεις στις χειρότερες ε, ανθρωπικές κρίσεις στον κόσμο. Προσπαθεί να βοηθήσει στην επιβίωση και στην ε, ε, βελτίωση της ζωής των ανθρώπων που πλήττονται από τις κρίσεις αυτές. Και θα ήθελα να αναφερθώ τώρα στο θέμα των ε, ενισχύσεων σε μετρητά. Πώς γίνεται αυτό στα πλαίσια των διεθνών μη οργανώσεων, θα αναφερθώ επίσης ε, στη σημασία του να δημιουργήσουμε νέα στοιχεία ε, κατόπιν έρευνας και θα δώσω το παράδειγμα του Πακιστάν και θα μιλήσω επίσης για τις προϋποθέσεις επιτυχίας ε, σε ό,τι αφορά τις μεταβιβάσεις χρημάτων σε μετρητά. Η συνάδελφος πραγματικά εξήγησε πολύ καλά το μηχανισμό σε ό,τι αφορά την ενίσχυση σε μετρητά ε, και υπάρχουν πάρα πολλά επιχειρήματα έτσι ώστε αυτοί, αυτά τα προγράμματα να επεκταθούν. Βεβαίως ε, αυτή η ανθρωπιστική ε, ενίσχυση μπορεί να είναι πιο γρήγορη, μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική χάρη στα μετρητά. Έχουμε λοιπόν και εμείς ένα φιλόδοξο στόχο. Είμαστε υπέρ του στόχου του ΕΚΟ για το 35% και θα πρέπει να υπάρξει μία ευθυγράμμιση αυτών των προγραμμάτων σε μετρητά με αυτά που αποφασίστηκαν στην Κωνσταντινούπολη στα πλαίσια της συμφωνίας. Βεβαίως ε, υπάρχει το θέμα των χρημάτων αυτών καθ' αλλά υπάρχει το θέμα της αξιοπρέπειας που ανέφερε η συνάδελφος. Τα χρήματα αυτά τα μετρητά δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους να κάνουν οι ίδιες επιλογές τους, να θέσουν τις προτεραιότητές τους Αντί να του δίνουμε εμεί αυτά που νομίζουμε ότι χρειάζονται, χρησιμοποιούν αυτοί τα μετρητά για να αγοράσουν αυτά που θεωρούν αυτοί ότι χρειάζονται με βάση τι συνθήκε τι οποίε ζουν. Είτε μιλάμε για στέγαση, είτε μιλάμε για εκπαίδευση και παιδεία. Είναι κάτι που μπορεί να επηρεάσει θετικά και την τοπική οικονομία και βεβαίω έχει ένα ε, πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Επ' αυτή τη ε, βάση η Επιτροπή μα έχει ένα στόχο το 25% τη ανθρωπιστική ενίσχυση ε, να ε, δίδεται μέσω ε, της μεταφοράς μετρητών ε, έως το 2020. Είμαστε στο 16% αυτή τη στιγμή, δηλαδή έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς τον στόχο αυτόν. Ε, αυτό έχει να συμπληρώσει το συνολικό στόχο της απάντησης στις ανθρωπιστικές κρίσεις εντός 72 ωρών τα μετρητά μας δίνουν τη δυνατότητα να είμαστε πιο γρήγοροι στην αντίδρασή μας και θέλουμε ακριβώς να πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Όπως ακούσατε ήδη, η τεχνολογία παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά την συνδρομή σε μετρητά. 75% των επιχειρήσεών μας ε, στις διάφορες χώρες θα πρέπει ως το 2020 να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα τεχνικά δηλαδή να ε, χορηγήσουν ενίσχυση σε μετρητά. Θα αναφερθώ ε, λεπτομερώς στη συνέχεια σε αυτό. Πώς λοιπόν θεσμοθετούμε, ε, πώς ε, η μεταφορά σε μετρητά θα μπορέσει να γίνει ε, κεντρικό στοιχείο της προσπάθειάς μας. Αφενός έχουμε έναν, ε, έναν φιλόδοξο βεβαίως συνολικό στόχο, αλλά χρειάζεται και να είμαστε πιο έτοιμοι να απαντήσουμε στις κρίσεις με μετρητά θα πρέπει να σκεφτούμε δηλαδή τις τεχνικές τις, ε, υποδομές που χρειάζονται. Θα πρέπει οι συνάδελφοι στι διάφορε χώρε να είναι εξοπλισμένοι έτσι ώστε να μπορούν να χορηγήσουν μετρητά. Και σε ό,τι αφορά τις ανάγκες υποδομές, τις ανάγκες τις τεχνολογικές ε, και τι ψηφιακέ πληρωμέ. ε, οι ψηφιακέ πληρωμές μάλλον παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο και χρειάζονται συμπράξει για να συμβεί αυτό. Δεν είμαστε εμείς εμπειρογνώμονε ε, σε ό,τι αφορά ε, τα κινητά χρήματα, τις ψηφιακές μεταφορές, τις ηλεκτρονικές μεταφορές. Βασιζόμαστε σε ιδιωτικό τομέα για τη δική του πραγματογνωμοσύνη. Μπορούμε βεβαίως μέσω των σχέσεων με τον ιδιωτικό τομέα να βελτιώσουμε ε, τη χορήγηση σε μετρητά, με τη Western Union, με τη Mastercard, ε, έτσι ώστε όταν προκύπτει μια επίγουσα κατάσταση να μπορούμε άμεσα ε, να ανεργοποιήσουμε τον μηχανισμό αυτό, ενώ όταν μιλάμε για ψηφιακή ετοιμότητα. Βεβαίως ε, πρόκειται για μια παρέμβαση η οποία αξιολογείται ε, ευρέω. Στην Επιτροπή μας εξετάζουμε τα στοιχεία, εξετάζουμε τα διάφορα αποτελέσματα, εξετάζουμε, παραδείγματος χάρη αυτή τη στιγμή, πώς τα μετρητά μπορούν να παίξουν ρόλο στην προστασία των γυναικών. Ε, για να προστατευτεί, προστατευτούν από ε, την ενδοκογενειακή βία, πώς μπορούν να παίξουν ρόλο τα ε, μετρητά σε ό,τι αφορά τα προγράμματα ε, σύντησης. Βασικές ανάγκες δηλαδή. Πρέπει να σκεφτούμε επίσης το, το ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται αυτή η πολιτική. Έχουμε θέσει σημαντικούς στόχους ε, πέρσι στη Συνόδο από τους δωρητές ε, που ήρθαν οι στόχοι αυτοί, αλλά πρέπει να βελτιωθεί η γνώση, να βελτιωθεί η όρεξη και η αποδοχή των μετρητών ως ένας αποτελεσματικός τρόπος ε, χορήγησης ανθρωπιστικής βοήθειας. Θα ήθελα τώρα να μιλήσω για τις, ε, την έρευνα και την ανάπτυξη που διενεργούμε. Εμείς ε, θέλουμε η ο προγραμματισμό μα να βασίζεται σε συγκεκριμένα δεδομένα, σε στοιχεία. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε τρόπο να είναι πιο γρήγορη και πιο αποτελεσματική η μέθοδο με την οποία ε, χορηγούμε τα μετρητά αυτά, ιδιαίτερα σε ψηφιακό επίπεδο όταν έχουμε μια επίγουσα κατάσταση. Υπάρχουν μια σειρά από προβλήματα που έχουν να κάνουν με το χρόνο που χρειαζόμαστε για να εντοπίσουμε ποιοι ε, είναι οι δικαιούχοι, ποιοι είναι αυτοί που χρειάζονται τα χρήματα αυτά, ποιοι είναι αυτοί που έχουν πληγεί ε, από μια καταστροφή. Στο Πακιστάν διαπιστώσαμε ότι χρειάζεται καμιά φορά ίσως και 40 μέρες όταν συλλέγουμε δηλαδή τα, τα δεδομένα πηγαίνοντας σπίτι με σπίτι ε, για να βρούμε ποιοι είναι οι, ε, οι δικαιούχοι. Έχουμε λοιπόν βρει ένα σύστημα για να πηγαίνουν τα πράγματα πιο γρήγορα. Να υπάρχει ένα πιο αυτοματοποιημένο σύστημα όπου ήδη έχουμε στοιχεία για τι πιο ευάλωτε ομάδε πληθυσμού. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά, λοιπόν, τα στοιχεία αυτά για να εντοπίσουμε και κάποιου άλλου ανθρώπου που οι οποίοι δεν έχουν ε, συμπεριληφθεί σε αυτού του καταλόγου. Υπάρχει μια ε, εταιρεία τεχνολογίας που λέγεται Σεγκόβια, η οποία μα βοηθάει ε, για την δημιουργία αυτών των δεδομένων και διαπιστώσαμε χάρη σε αυτές τις συμπράξεις, χάρη σε αυτή τη νέα καινοτόμα προσέγγιση, ότι μπορούσαμε να μειώσουμε διαδύο τον χρόνο παράδοσης της ενίσχυσης. Ε, είχαμε λοιπόν πραγματικές, ε, πραγματική πρόοδο αποτελεσματικότητα. Βεβαίω είναι πιλωτική αυτή η έρευνα, θα πρέπει να το ε, δοκιμάσουμε και αλλού, αλλά τα πρώτα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρα. Τώρα, οι τεχνολογικές καινοτομίες τις οποίες περιέγραψα σε ό,τι αφορά τα ψηφιακά χρήματα, τα κινητά χρήματα, τις προπληρωμένες κάρτες, αυτό εξαρτάται και από την κατάλληλη υποδομή. Υπάρχουν σειρά από πρωτοβουλίε σε ό,τι αφορά την ε, οικονομική συμπερίληψη, την ένταξη, την, ψηφιακή, ένταξη στην ψηφιακή οικονομία, αλλά διαπιστώνουμε ότι συχνά η ανθρωπιστική προοπτική ή εντό ενό ανθρωπιστικού πλαισίου, το ανθρωπιστικό πλαίσιο μάλλον δεν ε, υπάρχει σε αυτή την ανάλυση, απουσιάζει. Η ψηφιακή οικονομική ένταξη ε, θα πρέπει να λάβουν υπόψη μια κατάσταση ανθρωπιστικής ε, ανάγκης. Εδώ βλέπετε ε, σε αυτό το χάρτη που έχουμε τις μεγάλες ανθρωπιστικές κρίσεις. Από τις 50 περίπου σημαντικές ανθρωπιστικές κρίσεις είναι μόλις τέσσερις αυτές όπου μπορεί να λάβουν χώρα αυτές τις ψηφιακές μεταβιβάσει χρημάτων. Όταν λοιπόν χτυπάει η κρίση, είναι, δεν υπάρχει δυνατότητα να μεταβιβαστούν τα χρήματα αυτά, να δοθούν τα χρήματα αυτά ψηφιακά. Πρέπει να δοθεί, να δοθεί λοιπόν μεγαλύτερη έμφαση το ανθρωπιστικό σκέλο ε, σε ό,τι αφορά την ψηφιακή οικονομική συμπερίληψη και τη σχετική ατζέντα. Βλέπουμε ότι υπάρχει βεβαίω μεγάλη βούληση προ την κατεύθυνση αυτή και αυτό μα αρέσει και από την ΕΚΟ, υπάρχει πρόοδο ό,τι αφορά τι κριτέ γραμμέ ε, για τα μετρητά. Μια σειρά από δωρητέ επίση ε, έχουν δεσμευτεί κατά φιλόδοξο τρόπο μετά την Συνόδο Κορυφή. Ε, η Επιτροπή μα είναι έτοιμη να βοηθήσει όπου αυτό χρειαστεί. Ευχαριστώ. Merci, Ευχαριστώ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους που ενδεχομένως να θέλουν να παρέμβουν. Θα ξεκινήσω από τον κύριο, από την κυρία Γκερέρο μάλλον, τον κύριο Γκερέρο συγγνώμη, ο οποίος ασχολείται με την ανθρωπιστική ενίσχυση. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε να ευχαριστήσω ε, την Σάρα Τράουτμαν αλλά και την κυρία Γιαγιασίνγκε για τις ε, πληροφορίες που μας έδωσαν. Εγώ θυμάμαι ότι ε, στη Σύνοδο Κορυφή τη Κωνσταντινούπολη ένα από του μεγάλου στόχου ήταν ε, η τεχνολογική καινοτομία και το πώ αυτή μπορεί να βελτιώσει την χορήγηση ανθρωπιστική βοήθεια. Νομίζω ότι εδώ έχει σημειωθεί πρόοδο. Πριν από μερικέ εβδομάδε ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οργάνωσα, μάλλον συμμετείχα σε μια συνάντηση με εμπειρογνωμόνων σε διάφορους τομεί καινοτομία σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια. Ήταν, παρούσα, ήταν παρόμονα ο κ. Ντεμπράουερ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Βεβαίως ε, οι μεταφορές χρημάτων σε μετρητά αλλά και άλλα σημαντικά στοιχεία τεχνολογικού χαρακτήρα μπορούν ε, πραγματικά να βελτιώσουν την ανθρωπιστική βοήθεια. Βεβαίω, σήμερα επικεντρωνόμαστε ε, ακριβώς ε, ε, στην μεταφορά, στη μεταβίβαση μετρητών. Υπάρχει μια ευρύτερη συνειδητοποίηση ότι πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο πληρεί τρεις πολύ βασικές προϋποθέσεις που το καθιστούν ιδιαίτερα θετικό. Πρώτα απ' όλα, ο ίδιος ο δικαιούχος, αυτός που έχει την ανάγκη, είναι αυτός που αποφασίζει πώς θα δαπανίσει τα χρήματα αυτά. Για τη στέγαση, για τη σύντηση, ε, για την τεχνολογία. Ε, παίρνει ο ίδιος την απόφαση, εν περιπτώσει. Οι αναγκαιότητες λοιπόν δεν ορίζονται ε, δεν επιβάλλονται κατά κάποιο τρόπο στους δικαιούχους, οι ίδιοι ε, τις καθορίζουν. Ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι το στοιχείο της αξιοπρέπειας. Όταν δηλαδή κάποιος έχει τη δυνατότητα ο ίδιος να αποφασίσει, ακόμα και να αποφασίσει το ίδιο με αυτό που του έχουν προτείνει. Ε, το γεγονός ότι μπορεί ο ίδιος να το αποφασίσει είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο αξιοπρέπειας. Και το τρίτο είναι η αποτελεσματικότητα. Διότι έτσι εξοικονομούμε πόρους ενθαρρύνουμε την τοπική οικονομία Είναι μια σειρά από ζητήματα, όπως τόσο βελτιώνονται. Θα ήθελα να κάνω βεβαίως για τρία ερωτήματα και στις δύο μιλήτριες για την κυρία Τράουτμαν. Το ΕΚΟ αυτή τη στιγμή ε, αντιπροσωπεύει 35%, μάλλον 35% της ενίσχυσης μέσω του ΕΚΟ προέρχονται από μεταβάσεις ε, μετρητών. Τώρα άλλοι σημαντικοί δωρητές, μιλάω για τους μεγάλους δωρητές, έτσι, σε τι ποσοστά βρίσκονται σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια δηλαδή που χορηγείται μέσω μεταφοράς μετρητών. Ένα άλλο ερώτημα τώρα. Πώς ε, το πολιτιστικό στοιχείο, ε, η κουλτούρα που επικρατεί στη χώρα όπου ε, χορηγείται η βοήθεια, πώς αυτό επηρεάζει ε, τη δυνατότητα που έχουν οι δικαιούχοι εκεί να εκμεταλλευτούν τη δυνατότητα που του δίνεται. Ε, υπάρχουν κάποιες οικογενειακές δομές, ε, ε κάποιες ε, δομές φιλετικές που είναι τελώς διαφορετικές σε, στην Αφρική ή στην Κολομβία παραδείγματος χάρη. Αυτές οι, οι δομές λοιπόν οι οικογενειακές όπου κάποιος είναι κυρίαρχος στην οικογένεια. Μήπως δεν μας δίνει επαρκή εχέγγυα έτσι ώστε ε, να γνωρίζουμε ότι όντως ο δικαιούχο είναι αυτός ο οποίος αποφασίζει πώς θα τη τα χρήματά του. Ε, έχετε εντοπίσει τέτοιου προβλήματα στις ε, προσπάθειές σας και στις δράσεις σας. Βεβαίως υπάρχουν διαφορετικές, διαφορετικές κουλτούρες, ό,τι αφορά το πού θα δαπανίσει κάποιος τα χρήματα αυτά, πώς θα τα διαθέσει. Σε ό,τι αφορά τώρα το πού θα δαπανηθούν τα χρήματα αυτά, άλλο ένα ερώτημα. Η κυρία Τράουτμαν είπε ότι αυτά τα χρήματα δεν χρησιμεύουν για να αγοράσει κάποιος ε, ή να έχει πρόσβαση σε ε, υγειονομικές υπηρεσίες ή δεν θα έπρεπε βάση περιπτώσει. Στη συνέχεια όμως η κυρία Γιαγιασίνγκε αναφέρθηκε στην παιδεία. Δηλαδή πέρα από την αγορά προϊόντων για την αγορά υπηρεσιών ε, χρησιμοποιούνται αυτά τα μετρητά. Διότι αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει και κάποια προβλήματα. Φανταστείτε, μια ανθρωπιστική κρίση ε, μακράς διαρκείας. Ε, θα μπορούσε αυτό να είναι ένα κίνητρο ε, για τη δημιουργία ιδιωτικών εκπαιδευτικών συστημάτων ή ιδιωτικών συστημάτων περίθαλψης ε, και να δημιουργηθεί μια πελατεία μέσω αυτών των μετρητών που δίνουμε ως ανθρωπιστική βοήθεια. Ποια είναι η θέση σας επ' αυτού. Και κάτι ακόμα. Φαντάζομαι ότι σε πολλές περιπτώσεις έγινε αναφορά προηγουμένω στο Αφγανιστάν, αν κατάλαβα καλά, ε, όπου μπορεί να περάσουν εβδομάδες ως ε, του ε, κάποιος ε, εντοπιστεί και ταυτοποιηθεί ως δικαιούχος βοήθειας ε, Ορισμένε φορές φαντάζομαι ότι ακολουθείται ταυτόχρονα η διαδικασία της κλασικής ανθρωπιστικής βοήθειας ε, και η διαδικασία της ε, μεταβίβασης μετρητών. Μάλιστα, ευχαριστώ κύριε Γκερέρο. Άλλες παρεμβάσεις. Να δώσω το λόγο τις δύο εμπειρογνώμονες για να απαντήσουν στην, ε, στις ερωτήσεις του κ. Γκερέρο και στην παρέμβασή του. Ευχαριστώ πολύ τον ε, κύριο Κεραίρο για τις ε, πολύ καλές ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποιες από αυτές και να δώσω το λόγο και στη συναδελφό μου. Συμφωνώ απολύτως με την θέση σας όσον αφορά τη δυνατότητα να αποφασίζουν οι άνθρωποι οι ίδιοι τι θέλουν να κάνουν και από την άλλη να μην ε, σπαταλούν τα χρήματα που τους δόθηκαν. Αυτό είναι γενικά ο στόχος μας ε, που προσπαθούμε να πετύχουμε σε συνεργασία με τους εταίρους μας που παρέχουν τη βοήθεια. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ακόμα μαζί μας. Ελπίζουμε να συνεχίσει να συμμετέχει στην ε, προσπάθεια να παρέχουμε βοήθεια υπό τη μορφή μετρητών σε όλο τον κόσμο. Κάποιοι άλλοι από τους ε, μεγάλους δωρητές δεν ε, λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Ε, συνήθως διαθέτουν χρήματα για συγκεκριμένους στόχους. Αλλά στις συζητήσεις μας με τους διάφορους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών και με άλλους εταίρους ε, συχνά οι προτάσεις προέρχονται από τις ίδιες υπηρεσίε των Ηνωμένων Εθνών, τους ίδιους τους οργανισμούς. Ε, λένε ότι χρειαζόμαστε μετρητά, γιατί δεν μπορούμε να το ταιριάξουμε αυτό στην γενική μας προσέγγιση. Νομίζω ότι αυτό είναι ένας κοινό στόχος. Αλλά βέβαια όλα εξαρτώνται από το πόσο θέλουμε να σπρώξουμε την υπόθεση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται πολύ ψηλά όσον αφορά την επίτευξη των στόχων μας, ε, διότι έχουμε τις επιχειρήσεις αυτές ε, στην Τουρκία και αλλού όπου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το μέσο, ενώ σε μέρη όπως είναι η Σομαλία θα έχουμε γενικά ε, χαμηλότερο ποσό μετρητών που θα πρέπει να μοιραστεί σε περισσότερους ανθρώπους και τους εταίρους μας θα πρέπει να τους χρηματοδοτήσουμε όλους. Δεν μπορούμε να έχουμε λοιπόν ένα κεντρικό κανάλι παροχής μετρητών. Πιστεύουμε ότι ένα ποσοστό μέχρι 50% κάποια στιγμή είναι ρεαλιστικό. Κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά δεν νομίζουμε ότι πολλοί άλλοι δωρητές βρίσκονται στα ίδια επίπεδα με εμάς αυτή τη στιγμή όσον αφορά το πόση ελευθερία έχουν οι άνθρωποι για ε, να δαπανίσουν αυτά τα χρήματα και πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι τα χρήματα αυτά καταλήγουν ε, σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Γενικά, ε, ο στόχος μας είναι τα νοικοκυριά, όχι τα άτομα, διότι συνήθως υπάρχει κάποια οικογενειακή δομή την οποία δεν μπορούμε να παραβλέψουμε. Ο στόχος λοιπόν γενικά είναι το νοικοκυριό, αλλά δίνοντας τα χρήματα στη γυναίκα που είναι επικεφαλής του νοικοκυριού, νομίζουμε ότι αυξάνεται η πιθανότητα να χρησιμοποιηθούν με λογικό τρόπο τα χρήματα αυτά. Ε, με τις ε, πληρωμές σε μετρητά αποφεύγουμε κάποια από τα προβλήματα που έχουμε με άλλες μορφές βοήθειας. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις αυτό δεν ήταν δυνατό. Και επανέρχομαι σε αυτό που είπα νωρίτερα. Χρειαζόμαστε ένα ισχυρό πλαίσιο προστασίας ε, και όταν ε, δίνουμε βοήθεια σε μετρητά. Δεν ε, αρκεί απλά να βάζουμε μετρητά στο σύστημα. Ε, πολλές γυναίκες στη Μέση Ανατολή μας είπαν ότι προτιμούν να μην λαμβάνουν τη βοήθεια υπό μορφή μετρητών, διότι τίθεται θέμα ασφαλείας. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε άλλους τρόπους να διανύμουμε την βοήθεια. Ε, όπως είπε η συνάδελφος, είναι και ένας τρόπος να αντιμετωπίσουμε θέματα ισότητας των δύο φύλων, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε ώστε να μην χρησιμοποιήσουμε επιπλέον προβλήματα για τα κορίτσια και τις γυναίκες. Θα αφήσω τη συνάδελφό μου να απαντήσει. Έχω να κάνω και μια παρατήρηση όμως όσον αφορά τις ε, υπηρεσίες ε, εκπαίδευσης, αλλά θα επανέλθω σε αυτό. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικές. Θα ήθελα να πω λίγα πράγματα όσον αφορά τον ε, πολιτιστικό αντίκτυπο στις οικογένειες. Ένα θετικό παράδειγμα που είδαμε ήταν ότι οι οικογένειες μας είπαν ότι το να έχουν επιλογή σχετικά με το τι ε, τροφή θα αγοράσουν ε, έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην επιστροφή στην κανονικότητα. Να αγοράσουν δηλαδή το φαγητό που αρέσει στα παιδιά τους. δίδεται η δυνατότητα μεγαλύτερης ε, επικοινωνίας με την τοπική κοινότητα με τον τρόπο αυτό, όπως είδαμε και στην Ελλάδα. Ε, πιστεύουμε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Όσον αφορά την δυναμική εντός ε, της κάθε οικογένειας, θα συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε η συνάδελφος. Η ισότητα των φύλων και οι πιθανοί κίνδυνοι απασχολούν πολύ την Επιτροπή μας, την Διεθνή Επιτροπή Διάσωσης. Ε, εξετάζουμε λοιπόν τον ε, αντίκτυπο στην ε, δυναμική εντός της κάθε οικογένειας όταν δίνουμε μετρητά κατευθείαν στη γυναίκα. Γνωρίζουμε ότι αυτό μπορεί να γίνει με τρόπο πιο ασφαλή. Για παράδειγμα, να μην χρειάζεται να έρθει η γυναίκα να πάρει τα μετρητά, αλλά να γίνει η μεταφορά χρημάτων μέσω του κινητού τηλεφώνου. Εξετάζουμε λοιπόν ε, ποιος είναι ο αντίκτυπος ε, στην ε, δυναμική της οικογένειας καθώς και το πώς επηρεάζονται κορίτσια στην εφηβεία, πώς μπορούμε να τις ενδυναμώσουμε με πληρωμές σε μετρητά. Εξετάζουμε αν θα έχουν μεγαλύτερο ρόλο στην οικογένεια. Όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν προσπαθούμε να τα ε, συμπεριλάβουμε στον προγραμματισμό μας. Όσον αφορά την ερώτησή σας για την εκπαίδευση, νομίζω ότι πολύ σωστά το θίξατε αυτό. Εξετάζουμε τις δυνατότητες των ανθρώπων να δαπανίσουν τα χρήματα και ε, να έχουν ήδη άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες που ε, χρειάζονται, τι υπηρεσίες επιλέγουν. Εξετάζουμε τα θέματα αυτά όμως ε, κατά περίπτωση. Μία ακόμη παρατήρηση. Νομίζω επίσης ότι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι πληρωμές για τις οποίες ε, μιλάμε δεν θα επιτρέψουν σε κανένα να στείλει το παιδί σε ιδιωτικό σχολείο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια χρήματα για εκπαίδευση, αλλά αυτά καλύπτουν την ε, βασική εκπαίδευση. Δεν ε, θέλουμε ε, να χρεώνονται ξαφνικά τέλη για υπηρεσίες υγείας επειδή οι άνθρωποι θα έχουν χρήματα στα χέρια τους. Όπως είπε η συνάδελφος όμως ε, δίνουμε περιθώριο επιλογής στους ανθρώπους. Έτσι επιλέγουν οι ίδιοι και έτσι μπορούν πιο εύκολα να οργανώσουν τη ζωή τους. Ευχαριστώ. Merci, Ευχαριστώ κύριε. Πάμε τα σχόλια. Άλλες παρατηρήσεις. Ωραία. Ευχαριστούμε τις δύο εμπειρογνώμενους για την πληροφόρηση που μας παρέσχουν. Το επόμενο θέμα είναι η ψηφοφορία που προβλέπεται για τις 6 και 10. Οπότε είναι παρατέταρτο. Τελειώσαμε πιο σύντομα. Οπότε θα ξαναρχίσουμε στις 6 και 10. Ευχαριστώ πολύ.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

Chers collègues, si vous voulez bien prendre... Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Για να ψηφίσουμε. D'accord. On peut faire un essai sur... να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία για να δούμε αν λειτουργούν οι κάρτες σας. Άρχεται η ψηφοφορία.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 Σαμπάτου. Πέρας. Ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Τροπολογία 1. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αλλά ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Τροπολογία 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Νομίζω απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Donc le, le 3 il est... Le 4 était oui. D'accord, bon. Καλώς, καλώς, με συγχωρείτε. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές νομίζω απορρίπτεται να ελέγξουμε να ελέγξουμε άρχεται πέρας απορρίπτεται προφορική τροπολογία 1 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Α, θέλετε να ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 7 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Λοιπόν, τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω απορρίπτεται. Καλά να ελέγξουμε. Ελέγχουμε την τροπολογία 10 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 11. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε τροπολογία 9 τροπολογία 9 άρχεται πέρας εγκρίνεται τροπολογία 12 Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω εγκρίνεται. Εγκρίνεται, ωραία. Τροπολογία 14. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω εγκρίνεται. Οπότε περνάμε στη συμβαστική 2. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Οπότε περνάμε στο τροπολογία 23. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία. Προπολογία 29. Υπέρ. 29 λέω. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Να ελέγξουμε την 29 λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 30. Η τροπολογία 30 παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εάν εγκριθεί η προφορική τροπολογία 2, η τροπολογία 33 καταπίπτει. Λοιπόν, τροπολογία, προφορική τροπολογία 2, πρώτο τμήμα παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λοιπόν, καταπίπτει 33. Οπότε περνάμε στην τελική τελική ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται με 15 ψήφους υπέρ και μία κατά. Ωραία. Ε, euh, λοιπόν, συγγνώμη. Να ολοκληρώσουμε τη συνεδρίασή μας. Περνάμε στο σημείο 8. Ε, δεν υπάρχουν ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα περνάμε στο 9. Διάφορα. Δεν υπάρχουν διάφορα. Σημείο 10. Οι επόμενες συνεδριάσεις μας θα γίνουν στις 2 Οκτωβρίου τρέχοντος, στις 9 Οκτωβρίου τρέχοντος και τις 10 Οκτωβρίου τρέχοντος μηνός. Ε, έτους, συγγνώμη. Η συνεδρίασή μας ε, ολοκληρώνεται. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Σας εύχομαι καλό βράδυ και ευχαριστούμε για τις διερμηνείς. Oui, le vote, il est un peu chaotique.